πρακτικά θα τεθούν υπόψη του Κοινοβουλίου για έγκριση στην επόμενη ε, σύνοδο. Τα ψηφίσματα που επεγκρίθηκαν θα ε, διαβιβαστούν στα